Bien, nous allons commencer, ça va faire venir nos collègues. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε. Σήμερα έχουμε μαζί μας δύο ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε δύο τομείς που αποτελούν πηγή ικανοποίησης για μας. Έχουν να κάνουν με την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας στο επιχειρησιακό τμήμα, στο θεσμικό τμήμα. Και βέβαια θέλουμε success stories, θέλουμε δηλαδή επιτυχίες. Τώρα έτσι έχουμε στραμμένα τα μάτια πάνω το κεφάλι μας προς το διάστημα. Όταν πήγαμε στο Τορεχόν, κράτησα τις καλύτερες εντυπώσεις. Ήταν η πρώτη αποστολή της Επιτροπής μας, τη θητή αυτή, το 2009. Πήγαμε εκεί στο διαστημικό, στο κέντρο μάλλον δορυφόρων που έχουμε εκεί. Εκεί μας υποδέχτηκε ο κύριος Λοβρέντσιτς και θυμάμαι ότι αυτά που μας παρουσίασε τότε επιβεβαιώθηκαν στις επόμενες επισκέψεις που κάναμε στη συνέχεια επιτόπου σχετικά με τις αποστολές της κινήτησης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Γεωργία, για παράδειγμα, θυμάμαι την αποστολή μας στη Γεωργία, η οποία χρειάζεται δορυφορική απεικόνηση πάρα πολύ, όπως επίσης στην Αταλάντα που πήγαμε φέτος και είδαμε πώς χρησιμοποιείται και ποιοτικά και ποσοτικά πολύ ικανοποιητικά ε, το κέντρο. Εσείς θα μας πείτε βέβαια περισσότερα για την λειτουργία του κέντρου αυτού και για τις προοπτικές του. Θα μας μιλήσετε επίσης και για τους πόρους που διαθέτετε, τόσο οικονομικούς όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί και αυτό είναι χρήσιμο. Θέλουμε να το ξέρουμε. Και να μας πείτε επίσης πώς το κέντρο σας διαρθρώνεται με διάφορες αποστολές και μάλιστα και μελλοντικέ αποστολές και όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Φιλίπ Μπρουνέ που είναι διευθυντής για την ε, αεροδιαστημική βιομηχανία μέχρι τώρα, χτυπάμε ξύλο βέβαια, έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή διάρθρωση στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα. Κάτι το οποίο εμεί θέλουμε από τη δικιά μας τη θέση, δηλαδή αυτό ζητάμε. Έτσι ώστε η επιχειρησιακή διάσταση και αν πρέπει και στρατιωτική να υπάρχουν και να υπάρχει καλή συνεργασία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε να επωφεληθούμε για τις αποστολές της κοινή πολιτικής ασφαλής και άμυνας δώσει και αυτό με το πρόγραμμα Κοπέρνικους ή το άλλο εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για τον γεωπολιτικό εντοπισμό, το Γαλιλαίο. Και έχουμε βέβαια και όλες τις συζητήσεις που γίνονται στον τομέα της έρευνας που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της διαδικασίας που θα καλύψει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Ο κύριος Μπρουνέ συμμετείχε πάρα πολύ στην προετοιμασία του τρίτου καλαθιού για τη βιομηχανία μετά από την ανακοίνωση των Επιτρόπων Μπαρνιέ και Ταγιάννη που ήρθαν και μας εξήγησαν εξάλλου. Συνεπώς εδώ βλέπουμε να υπάρχουν ενδιαφέρουσες προοπτικές. Ότι υπάρχει άνοιγμα και ότι αν έχουμε επιτυχίες σίγουρα το διάστημα δεν θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα έχουμε τις επιτυχίες αυτές. Κάθε άλλο. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε και θέλω να σας δώσω το λόγο. Πρώτα στον κύριο Μπρουνέ ίσως. Σύμφωνε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τανζάν. Θα προσπαθήσω σύντομα, πριν ακριβώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, να σας αναφέρω το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και βρίσκεται το διάστημα στις συζητήσεις δηλαδή που γίνονται όσον αφορά την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Όπως το υπενθυμίσατε κι εσείς, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό γιατί, γιατί έχει στατικής σημασίας ενδιαφέρον για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί χωρίς το διάστημα δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε σωστές αποφάσεις, το σχεδιασμό και τις δράσεις για να ανταποκριθούμε στην κρίση. Είναι αλήθεια βέβαια ότι έχουμε ήδη κάποιες επιτυχίες. Η διαστημική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, είναι πρόσφατη, γιατί διευκρινίστηκε με ανακοίνωση το 2011 μόνο. Επί τη ευκαιρία της ανακοίνωσης αυτής διευκρινίσαμε τότε τις διάφορες πλευρές της διαστημικής πολιτικής που θέλει να δώσει απαντήσεις σε προκλήσεις της κοινωνίας, δημόσια ασφάλεια, ασφάλεια των πολιτών, ανθρωπιστικά μεταφορές, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν και προκλήσεις οικονομικές και το διάστημα μπορεί να βοηθήσει. Γιατί, γιατί μας βοηθάει με γνώση. Είναι μια όθεση που παίρνουμε στις τεχνολογίες εχμής. Επίσης, δημιουργεί θέσει απασχόληση στο διάστημα. Και έπειτα πρόκειται και για μια πρόκληση στρατηγική σημασία, όπω είπατε και εσεί, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει τη θέση που τη πρέπει στον κόσμο χωρί το διάστημα. Δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη οικονομικά και πολιτικά χωρί να έχει τα ατού, τα διαστημικά που έχουν οι άλλε μεγάλε δυνάμει. Αναφερθήκατε και σας ευχαριστώ για αυτό στους δύο πυλώνες που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων πρωτοβουλειών δηλαδή θα μας επιτρέψουν και δύο αυτοί πυλώνες να πετύχουμε τους στόχους μας. Πρόκειται για το Κοπέρνικο και το Γαλιλαίο. Πρώτον, τα δύο αυτά εργαλεία είναι μη στρατιωτική υποδομή υπό έλεγχο μη στρατιωτικό. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί συχνά κάνουμε την σύνδεση με άλλες παρόμοιες δομές και εκεί είμαστε αντιμέτωποι με στρατιωτικές δομές ή μικτές υποστρατιωτικό έλεγχο και όχι τόσο μη στρατιωτικές. Στην Ευρώπη όμως φτιάξαμε αυτό το σύστημα δεχόμενοι ότι οι υποδομές αυτές, ακριβώς επειδή είναι μη στρατιωτικού χαρακτήρα, μπορούν να εξυπηρετήσουν και τους χρήστες της άμυνας με τη βοήθεια δορυφόρων, ε, ε, τηλεπικοινωνιών, εμπορικών ή να εξυπηρετήσουν και άλλες εφαρμογές και άλλα προϊόντα όπως είναι το HumetSat. Θα αναφερθώ τώρα στις διάφορες αυτές δομές. Πρώτα απ' όλα για το Γαλιλαίο. Είχαμε την πρώτη αυτόνομη τοποθέτηση του συστήματος τον Μάρτιο του 2013 και ιδιαίτερα το σύστημα PRS που είναι οι υπηρεσίες υπό κρατικό έλεγχο γίνονται πια πραγματικότητα. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό. Διότι το σύστημα αυτό του Γαλιλαίου, η κρατικά ελεγχόμενη υπηρεσία δηλαδή, θα προσφέρει συνέχεια υπηρεσιών κάτι το οποίο δεν διασφαλίζει σήμερα το GPS, το σημερινό σύστημα. Ακόμα δηλαδή και σε περιπτώσεις κρίσεων των πιο μεγάλων, αυτό το σύστημα θα συνεχίσει να λειτουργεί και δεν θα επηρεάζεται από προσπάθειες παρεμβολών. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν εννοείται ότι είναι μια επιλογή για όλες τις δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη διατήρηση της τάξης, όπως επίσης και με δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την άμυνα στα κράτη-μέλη. Σήμερα Υπάρχει μια πράξη που εξετάζει τώρα το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να έχουμε ελάχιστε κοινέ προδιαγραφέ που θα εφαρμόζουν οι χώρε μέλη. Γιατί είναι βέβαιο, όπω καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικό όλε οι χώρε μέλη που στο μέλλον θα χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε αυτέ να μπορούν να έχουν κοινέ προδιαγραφέ, ώστε να λειτουργούν συντονισμένα. Και γιατί το λέω αυτό, πιο συγκεκριμένα το λέω, γιατί πρόκειται για κατεξουσιοδότηση πράξη Οπότε εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε μια θετική επιρροή. Εξαρτάται δηλαδή από το κατά πόσο γρήγορα θα εγκριθεί αυτή η ή πράξη για να προχωρήσουμε. Έρχομαι τώρα στον Κοπέρνικο. Να σας πω εδώ δύο λόγια για το τι είναι ο Κοπέρνικος. Ο Κοπέρνικος είναι μια υπηρεσία με τρεις συνιστώσεις. Μια συνιστώσα υπηρεσίες, μία συνιστόσα δορυφόρη και μία συνιστόσα με αισθητήρε ε, in situ το Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο Κοπέρνικος, ενώ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα δορυφόρο, εδώ και πολλά χρόνια έχει αρχίσει να λειτουργεί και μάλιστα λειτουργεί εύρυθμα. Αν δεν το σημειώσετε. Ε, δεν πειράζει, σας το λέω τώρα. Ο πρώτος χάρτης που κυκλοφόρησε παγκοσμίω μετά τη, το τυφώνα Γιάννα στις Φιλιππίνες ήταν ένας χάρτης ε, που προήλθε από το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Ε, τώρα, η διαστημική συνιστόσα είναι έξι οικογένειες από δορυφόρους Sentinel. Έξι δηλαδή οικογένειες δορυφόρων που ο καθένας θα δώσει διαφορετικά είδη δεδομένων. Για κάθε οικογένεια δορυφόρων ε, θα υπάρξει και συνέχεια. Ο πρώτος ε, Sentinel θα ξεκινήσει από τη βάση εκτόξευσης ε, στο Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας τον Απρίλιο του 2014 και θα εκτοξευθεί με πύραυλο Σογιούς. Αλλά έχουν προβλεφθεί και άλλοι δορυφόροι αργότερα για το 2014 ο Sentinel-2 και ο Sentinel-3. Ο Sentinel-1 είναι ραντάρ, ο δεύτερος δορυφόρος είναι οπτικός και ο τρίτος δορυφόρος Sentinel είναι μικτός δορυφόρος, δηλαδή περιέχει δελτίμετρα και επίση κάποια στοιχεία εδαφικά. Στο όλο αυτό αρχιτεκτόνημα θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχουμε και κάποια συμμετοχή ε, των κρατών μελών στις αποστολές. Γιατί δεν έχουμε δορυφόρους υψηλή ευκρίνεια ε, που να προβλέπονται στο Κοπέρνικο, αλλά κάποια κράτη-μέλη που ήδη έχουν τέτοιου δορυφόρου ε, υψηλή ευκρίνεια συμμετέχουν, συμβάλλουν σε αποστολέ. Και σε τέτοιου είδου αποστολέ ε, λαμβάνουμε στοιχεία και μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου χάρτε όπω αυτό που σα ανέφερα. Τρει έχουμε τέτοιε κοινέ αποστολέ με τη Γαλλία στον αστερισμό Πλεάδες, ε, με τη Γερμανία για την ε, ε, Γερμανία στο Τέρα Αρίξ και για την Ιταλία στο Κόσμο Sky. Και μια και εδώ έχουμε την υποεπιτροπή σας που ασχολείται με την άμυνα. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση αυτά τα στοιχεία που δίνουν τα κράτη-μέλη σε αυτές τις κοινέ αποστολές, έχουμε κάποια στοιχεία υψηλής ευκρίνειας που συνδυάζονται με τα στοιχεία του Κοπέρνικος και που δεν είναι διαθέσιμα γιατί ε, μόνο τα κράτη-μέλη έχουν δεδομένα υψηλή ευκρίνηση. Χάρη σε αυτόν τον συνδυασμό δίνουμε σημαντική προστιθέμενη αξία σε δραστηριότητες άμυνας και ασφάλειας. Το GMES ήταν ο πρόδρομος του Κοπένικου. Στο S, ε, στο ακρόνιμο, ε, αντιστοιχεί στην ασφάλεια. Και εκτός από τους χάρτες που σας είπα ε, που έγινε μετά τον κυκλώνα στις Φιλιππίνες, έχουμε τρεις τέτοιες υπηρεσίες. Η πρώτη υπηρεσία του Κοπέρνικους ε, προσφέρει στήριξη στην επιτήρηση των συνόρων, είναι η πιο προηγμένη και με τον κανονισμό Eurosur που θα τεθεί σε εφαρμογή καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που λένε η στρατηγική κονόψα, αρχική ιδέα ενέργειας των επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την επιτήρηση και των χερσαίων και των θαλάσσιων συνόρων ε, στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη με βάση ε, κοινά διαστημικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε από διάφορες πηγές πληροφοριών. Και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο σημαντικό. Το σύστημα Κοπέρνικος είναι ένα σύστημα που θα επιτρέψει την ε, ε συμπερίληψη και διασταύρωση στοιχείων από πολλές πηγές και διάφορες κατηγορίες ε, πληροφοριών. Σας μίλησα για το ραντάρ, το δελτιμετρία. Ε, θα έχουμε αισθητήρε επιτόπου, οπότε το τελικό προϊόν δεν θα είναι το απλό άθροισμα κάποιων στοιχείων αγοράς, αλλά θα είναι το άθροισμα μιας διασταύρωσης πολλών στοιχείων. Εκτός από τη στήριξη στην επιτήρηση των συνόρων, προσφέρουμε υπηρεσίες ε, για τις εξωτερικές δράσεις, ε, στήριξη των εξωτερικών δράσεων κάτι που ανταποκρίνεται στην ανάγκη της ΚΕΠΑ και της ΚΠΑ. Και εκεί χρησιμοποίησαμε διάφορα σενάρια σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την ΕΙΕΘ, που θα είναι φυσικά από τους σημαντικότερους χρήστες αυτών των επιχειρήσεων. Και μια και το Κοπέρνικος είναι ένα σύστημα που θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών, Συνεργαστήκαμε με την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με, την, ε, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Διαστήματος για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά της τη διαστημικής συνιστώσης του Κοπέρνικου για να ανταποκριθούμε ακριβώς στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Και σε ό,τι φορά τις ε, προθεσμίες απόκτησης που είναι σημαντικό και το ε, τις προθεσμίες νέων επισκέψεων. Δηλαδή πόσες φορές περνάει από το ίδιο σημείο ε, της γης ο δορυφόρος. Επίσης έχουμε και υπηρεσία θαλάσσιας επιτήρησης, πολύ γνωστή υπηρεσία που υπάρχει ήδη σε διάφορες χώρες μέλη και το σύστημα Κοπέρνικος θα συμπληρώσει τις ε, υπάρχουσες υπηρεσίες θαλάσσιας επιτήρησης και θα πρέπει βέβαια να προσδιορίσουμε καλύτερα κάποια στοιχεία τη διακυβέρνηση του συνόλου αυτών των υπηρεσιών θαλάσσια επιτήρηση. Ο πρόεδρο ο κ. Ντανζόν, αναφέρθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Άμυνα. Εγώ θα σας αναφέρω ένα άλλο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είχε αποφαστεί περίπου την ίδια εποχή, το Φεβράριο του 2013, αλλά η προετοιμασία είχε γίνει από το Δεκέμβριο του 2012 και προς έκπληξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επανένταξε το Κοπέρνικο στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάτι που οδήγησε σε κάποιες αναπροσαρμογές της στρατηγική γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ως νομική βάση για το σύνολο των σημείων που είχε ίδια συμπεριλάβει στο πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί δεν υπήρχε το Κοπέρνικος εκεί και δεν υπήρχε νομική βάση. Μετά την ένταξη του Κοπέρνικου στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χρειάστηκε μία νομική βάση. Έχουμε ζητήσει λοιπόν μια νομική βάση για το Κοπέρνικος και ελπίζουμε ε, στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να διεκπεριωθούν εγκαίρως οι προετοιμασίες κατά το πρώτο εξάμεινο του 2014, ώστε, και εδώ θα ήθελα να είμαι σαφής και κατηγορηματικός γιατί ενδιαφέρει αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ελέγχει το πρόγραμμα, αλλά ενδιαφέρει και όλους τους οικονομικούς τελεστές, τα θεσμικά όργανα, τα τους φορείς στα κράτη-μέλη που θα χρησιμοποιήσουν και θα συνεργαστούν με το Κοπέρνικους για να εξασφαλίσουμε την ε, εκτέλεση του προπολογισμού του Κοπέρνικους για το 2014 θα πρέπει προηγουμένω να έχουμε μια σταθερή νομική βάση ήδη από το 2014 διαφορετικά και η βιομηχανία και ε, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματο θα χάσουν 430 εκατομμύρια ευρώ για το 2014. Δεν είναι μόνο θέμα προθεσμίας, δηλαδή είναι ότι δεν θα μπορέσουν να εκταμιευθούν τα κονδύλια που προβλέπονται για το Κοπέρνικου ε, για το 2014, γιατί δεν έχουμε την νομική βάση, δεν θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε καταξιοδότηση πράξη και άρα δεν θα μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε αυτό το κονδύλιο. Επίσης, άλλο σημαντικό θέμα του Κοπέρνικους είναι η πολιτική των δεδομένων, ένα αναπόσπαστο στοιχείο του Κοπέρνικου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Ιουλίου πέρυσι ενέκρινε ε, έναν κανονισμό που είναι κατεξουσιοδότηση πράξη, χωρίς αντιρρήσεις ε, από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα τεθεί ε, σε ισχύ σε 9 Δεκεμβρίου. Και αυτό το κείμενο, αυτός ο κανονισμός προσδιορίζει τις προϋποθέσεις για μια πλήρη ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση του τέστην, όλες οι εμπορικές εφαρμογές θα είναι δυνατές, εφικτές, με βάση τα δεδομένα που προσφέρονται από το Κοπέρνικος, από το σύστημα αυτό. Και η μελέτη επιπτώσεων ε, που συνόδευσε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσδιορίσε 48.000 χρήσεις και, 30, ε, και θέσεις απασχόλησης και 30 ε, δισεκατομμύρια ευρώ κυκλοργασιών για την περίοδο αναφοράς την περίοδο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Βέβαια, επειδή έχουμε ανταγωνισμό με τους Αμερικανούς ε, με το δικό του σύστημα σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ανοιχτή και δωρεάν πρόσβαση, με αυτή την πολιτική των δεδομένων θα έχουμε πολύ θετικά στοιχεία και πολλά οικονομικά ωφέλη από το Κοπέρνικος. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή για μια παρατήρηση στη συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο για τα δεδομένα του Κοπέρνικος. Πολλοί αναφέρθηκαν στο θέμα της ασφάλειας. Δεν ξέρω πώς θα, θα εξελιχθεί η συζήτηση, γιατί ο σχετικός κανονισμός για το Κοπέρνικος δεν έχει ακόμη εγκριθεί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση, αλλά όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, το σύστημα Κοπέρνικος έχει στο DNA του, στα γονίδια του, το πολιτικό σκέλος, μη στρατιωτικό. Και από την ίδια την ύπαρξή του εκφύσεως και από τα δεδομένα του θα βοηθήσει κυρίως την ασφάλεια και την άμυνα. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτό το στάδιο να ζητήσουμε από το Κοπέρνικος να γίνει ένα σύστημα ασφάλειας και άμυνας. Δηλαδή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε στο Κοπέρνικο και στους δορυφόρους του ιδιαίτερος μια πολιτική δεδομένων ε, για την οποία δεν είχαν να σχεδιαστεί. Για παράδειγμα, έχουμε τους δορυφόρους τους ΜΕΤΣΑΤ με τα μετεωρολογικά στοιχεία που είναι ε, εξαιρετική σημασίας για την άμυνα. Αλλά οι, αυτοί οι μετεωρολογικοί δορυφόροι δεν είχαν κατασκευαστεί για την άμυνα. Οπότε 80% ε, των πολιτικών εφαρμογών, αν το σύστημα μετατραπεί σε στρατιωτικό, θα εξαφανιστούν. Τώρα, αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Σύμβουλο που κατά πάσα πιθανότητα θα σχολιάσει τα δύο συστήματα, το Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικο. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα τρίτο σύστημα το σύστημα που αφορά την αποκατάσταση ασφάλειας στο διάστημα. Δηλαδή, πρόκειται για διαστημικές υποδομές και προκειμένου τους δορυφόρους. Εδώ πρέπει να ομολογήσουμε την σημαντική μας και αυξανόμενη μάλιστα εξάρτησή μας από τις υπηρεσίες τρίτων χωρών. Έχουμε και δικές μας διαστημικές υποδομές. Αλλά για να εξασφαλίσουμε τη συντήρησή τους και τη διάρκεια τους, εξαρτόμαστε από υπηρεσίες που δεν είναι ευρωπαϊκές. Εξαρτόμαστε δηλαδή από τρίτους. Μία από τις σημαντικές απειλές είναι τα θράψματα και τα διαστημικά απόβλητα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τι είναι αυτά τα διαστημικά απόβλητα. Δεν ξέρω αν είδατε την ταινία Gravity Αυτά τα διαστημικά απόβλητα, τα διαστημικά σκουπίδια είναι τεράστια απειλή γιατί πρόκειται για θράσματα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη τροχιά και απειλούν τους δορυφόρους. Και στα πλαίσια του ορίζοντα 2020 έχουμε κάποια σχέδια για να αποφύγουμε την, τον πολλαπλασιασμό τέτοιων διαστημικών σκουπιδιών και έχουμε και ένα σύστημα για να καθαρίσουμε κατά κάποιο τρόπο συγκεκριμένες τροχές, αλλά αυτό το σύστημα που έχουμε είναι το κυρίως το σύστημα της αποφυγής. Οπότε για να αποφύγουμε ένα διαστημικό σκουπίδι πρέπει να ξέρουμε πού βρίσκεται για να δούμε πώς θα κινηθεί ο δορυφόρος. Μόνο την αποφυγή έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αλλά σε ένα τέτοιο περιβάλλον με τόσα πολλά διαστημικά σκουπίδια δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε ζωή τους δορυφόρου μας αν δεν έχουμε στοιχεία από τους Αμερικανούς. Έχουμε κάποιες ικανότητες και προτείναμε μάλιστα στην Ευρώπη ένα σύστημα στήριξης ε, για την επιτήρηση του διαστήματος και την παρακολούθηση ε, αντικειμένων ε, τροχιά. Είναι το SST, το σύστημα παρακολούθησης και χνηλάτησης εντοπισμού του διαστήματος και μάλιστα ε, σας ευχαριστούμε θερμά γιατί στηρίξατε την πρωτοβουλία μας και είναι σημαντικό ο Κοπέρνικος, παρά, παρόλο που δεν έχει τις ίδιες ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις, είναι σημαντικό αυτό το σύστημα το SST να τεθεί σε εφαρμογή πριν το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας. Και είναι μια έκκληση που θα ήθελα να απευθύνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως κάναμε και στο Συμβούλιο, να μεριμνήσει ώστε η διαδικασία έγκρισης για το SST να ολοκληρωθεί πριν τον Απρίλιο του επόμενου έτους. Και είναι προφανές ότι το Κοπέρνικος πολύ περισσότερο από το Γαλιλαίο ε, λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές στρατιωτικές ανάγκες από το σύστημα παρακολούθησης και εχνηλάτησης του διαστήματος. Γιατί ο εντοπισμός των ε, διαστημικών σκουπιδιών βέβαια βρίσκεται στα χέρια των στρατιωτικών. Αυτό ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να παρεύει στο ποιο κάνει τι. Το μόνο μας ε, σύνθημα, η μόνη αρχή στην πρωτοβουλία μας είναι ότι ε, θα πρέπει να βάλουμε σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο, να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν, ώστε να δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα. Και από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η σωστή δικτύωση, θα δούμε πώς θα αυξήσουμε τις ικανότητές μας, θα τις επικαιροποιήσουμε, ώστε κάποια στιγμή αργότερα, στο μέλλον, να έχουμε και ποιοτικά και ποσοτικά μια κρίσιμη μάζα, ώστε να μπορούμε να μιλούμε επίση ώρες με τους Αμερικανούς για να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερο συντονισμό. Αυτά προς το παρόν, ίσως στη συνέχεια με τις ερωτήσεις συμπληρώσω κάποια θέματα. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι στα πλαίσια των πιθανών συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κατά τη γνώμη μας, τρεις είναι οι σημαντικές πρόοδοι που θα μπορούσαν να γίνουν στα θέματα του διαστήματος. Πρώτον, πέραν των εφαρμογών του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου. δεν θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα, περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μία δέσμευση, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα να αναλάβουν δεσμεύσεις για να υλοποιήσουν αυτό το σύστημα παρακολούθησης και εχνηλάτησης του διαστήματος του SST. Επίσης το, σύστημα, το θέμα των επικοινωνιών ε, με δορυφόρους και το ελεύθερο αποτέλεσμα λόγω του κατακαιρματισμού της ζήτησης και εξαιτία των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων υπάρχουν και αφιβολίες για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς δορυφόρων των επικοινωνιών κυβερνητικών δορυφόρων. Και θα πρέπει λοιπόν ε, να συνεργαστούμε για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας και ενδεχομένως να υιοθετήσουμε κάποιες κοινέ στρατηγικές. Και τρίτο σημείο, το τρίτο που περιμένουμε από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, είναι το θέμα των δορυφόρων υψηλής ευκρίνειας και των της να αναπτύξουμε στρατηγικά νέες δυνατότητες απεικόνησης υψηλής ευκρίνειας για να καλύψουμε τις ανάγκες και ΠΑ και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι και η ΕΕΘ αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος θα πρέπει να αναμειχθούν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Εντάξει, λεπτομέρειε. Μετά θα σας τις θέσω. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Λεφρέντσης του κέντρου διαστήματος. Έχετε και slides, ε, διαφάνειες. Ωραία, οπότε θα πάμε και εμείς απέναντι για να μπορούμε να τις βλέπουμε καλύτερα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι μου δίνετε τη δυνατότητα να ξανάρθω στην Υποπιτροπή για Ασφάλεια και Άμυνα για να μπορέσω να σας ενημερώσω για το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μέσα στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται για το διάστημα και την ΚΠΑ. Χαιρόμαστε λοιπόν που μας προσφέρει την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα επιτεύγματα αυτής της, αυτού του γραφείου, αυτού του οργανισμού κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά επίσης ε, να καταδείξουμε και πώς μπορεί να υπάρξει πρόοδος ε, στο μέλλον. Η Υποεπιτροπή, το Κοινοβούλιο και όλοι οι θεσμοί που ασχολούνται με την ΚΠΑ και την ΚΕΠΑ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά το δορυφορικό κέντρο, θέλω να σας πω ότι έχουμε εδώ έναν θεσμό, έναν οργανισμό, ο οποίος λειτουργεί ως ε, οργανισμός του Συμβουλίου και έχει κατορθώσει να αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με τα κράτη-μέλη, κυρίως το χώρο που καλύπτει. Αναφέρομαι στην υποστήριξη της ΚΠΑ, της ΚΕΠΑ, και η αποστολή του δορυφορικού κέντρου δεν είναι απλά να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στην ανάλυση απεικονίσεων δορυφορικών, αλλά να βοηθάει και στην χάραξη πολιτικής. Θέλω αυτό να το υπογραμμίσω ευθύς εξ αρχής, διότι μερικές φορές η όλη συζήτηση για τη χρήση του χώρου ε, σταματάει μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό ε, σημείο που είναι τα τελευταία χιλιόμετρα μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εμείς στο δορυφορικό κέντρο τα τελευταία χρόνια καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για να καλύψουμε ε, να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει όσων χρησιμοποιούν το δορυφορικό κέντρο, ε, να τους ευχαριστήσουμε με βάση αυτά που υπάρχουν σε σχέση με το διάστημα. Η αποστολή του δορυφορικού κέντρου συζητιέται αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη και αναμένουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου ε, σύντομα για το δορυφορικό κέντρο. Ένα θέμα λοιπόν που συζητείται είναι ακριβώς πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση του διαστήματος δεν σταματάει απλά και μόνο ε, προσφέροντας ε, εντυπωσιακά προϊόντα, τα οποία όμως κάπου βρίσκονται και δεν ε, χρησιμοποιούνται κατά τη χάραξη μιας συγκεκριμένη πολιτικής. Θέλω λοιπόν αυτά κάπως να τα συζητήσουμε αν θέλετε κι εσείς. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι για να είναι κανείς επιτυχής σε, μια, σε ένα λειτουργικό φορέα όπως είμαστε εμείς πρέπει να ορίσει τη μορφή της ε, διαχείρισης που επιτρέπει στο κέντρο να στιαστεί στην αποστολή του. Οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τους ε, τομείς ενδιαφέροντος αυτό παραμένει ε, καθαρά στους πολιτικούς. Αναφέρομαι την ε, λειτουργική κατεύθυνση που χαράσει η ύπατη εκπρόσωπο και βεβαίω και τα κράτη-μέλη έχουν την εποπτεία. Αυτός ο τρόπος εργασίας έχει ενισχύσει την ε, νομοποίηση του κέντρου και Παρότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, θα ήθελα παρόλα αυτά να υπογραμμίσω τη σημασία αυτής της ε, νομιμοποίησης. Επίσης, θα ήθελα να υπογραμμίσω και τη σημασία των άμεσων ε, σχέσεων ε, των, των, το πόσο σημαντικό είναι να καθορίζουμε προτεραιότητες. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όσους χρησιμοποιούν το κέντρο. Θα αναφερθώ ε, σε αυτό αργότερα. Ε, ο πρόεδρος πολύ σωστά μίλησε προηγουμένως για αποστολές και επιχειρήσεις. Αν δει κανεί ε, το οργανόγραμμα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, το διαστημικό κέντρο εμφανίζεται σε αυτή την απεικόνηση. Βέβαια το κέντρο αυτό εξακολουθεί να είναι μια υπηρεσία του Συμβουλίου με επικεφαλής από την νομική υπηρεσία Βλέπουμε βέβαια ότι επειδή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης έχει πλέον ε, ε, θεσμοθετηθεί, αυξάνονται όλο και περισσότερο τα αιτήματα που καταλήγουν σε εμά για να ικανοποιήσουμε. Και προσπαθούμε όλα αυτά να τα ελέγχουμε, ε, να τα ικανοποιούμε με βάση τις πηγές που έχουμε. Το δορυφορικό μας κέντρο έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χρησιμοποιεί τόσο εμπορικές απεικονίσεις όσο και ε, κρατικές, κυβερνητικές. Στο εμπορικό επίπεδο σήμερα οι πιο σημαντικές πηγές ε, προέρχονται από την Ευρώπη. Αυτό νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο ε, γιατί επιθυμούμε ε, να έχουμε όλο και μεγαλύτερο ευρωπαϊκή αυτονομία. Εκτός λοιπόν από τους ε, εμπορικούς δορυφόρους, το δορυφορικό κέντρο χρησιμοποιεί και κυβερνητικούς πόρους από τρεις χώρες, από τη Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα, από το κόσμο SkyMed, ένα διτό σύστημα της Ιταλίας και από το σύστημα Σαλούπε της Γερμανίας. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει συνδυασμός των εμπορικών και των κυβερνητικών στοιχείων και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε πολύ εκλεπτισμένα στοιχεία που προσφέρουμε στους χρήστες μας. Επίσης μπορούμε να έχουμε και ευελιξία όσον αφορά την ταχύτητα προσφοράς των υπηρεσιών μας. Βεβαίως ε, υπάρχει και το αίτημα πολλές φορές ε, να μεταφέρει πληροφορίες σε ένα ευρύτερο φάσμα χρηστών, αλλά αντιμετωπίζουμε και πολύ συγκεκριμένα θέματα όπου οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες είναι πολύ περιορισμένοι. Ένας από τους τομείς όπου το δορυφορικό κέντρο αντιμετωπίζει δυσκολίες είναι όσον αφορά το υψηλότερο επίπεδο ευρωπαϊκής αυτονομίας. Πριν από κάποια χρόνια αγοράσαμε το 80% των δεδομένων, αγοράζαμε τα δεδομένα από την Αμερική και από άλλους μη Ευρωπαίους παρόχους. Και με χαρά μπορώ να σας πω ότι φέτος δεν επιτύχαμε πλήρη αυτονομία, αλλά εν πάση περιπτώσει το 60% των δεδομένων μας έρχονται από την Ευρώπη, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να αναφέρω το πόσο σημαντική είναι αυτή η ευρωπαϊκή αυτονομία ε, στον τομέα ε, των ε, εμπορικών απεικονίσεων υψηλής ευκρίνειας. Τα δεδομένα που αναλύουμε είναι πολλά και αυτό είναι απαραίτητο γιατί έχουμε και πάρα πολλούς χρήστες που μας αναθέτουν μια αποστολή. Το Intel Cycle, ο κύκλος αυτός μέσα στον οποίο δουλεύουμε, αποτελείται από διάφορους και διαφορετικούς χρήστες, από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, από αποστολές, ε, επιτόπου ελέγχους, ε, αλλά από το Incent, το CPPC, στρατιωτικούς συνεργάτες και άλλους. Πρόσφατα υπήρξε σημαντική αύξηση του αριθμού ετοιμάτων από έξω ευρωπαϊκούς θεσμούς, κυρίως από τα Ενωμένα Έθνη. Και Επίσης και μαζί σε δεδομένα και υπηρεσία για την απαγόρευση χημικών όπλων και θα αναφέρω αργότερα παραδείγματα. Ε, έχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους χρήστες και συνεχίζουμε την πολιτική μας που είναι ο έλεγχος της διαφάνειας σε σχέση με όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή όλες οι πολιτικές και τα προϊόντα μας προσφέρονται σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη να είναι ανα πάσα ώρα και στιγμή ενημερωμένα για το τι ακριβώς πράττουμε. Όσον αφορά τώρα τα προϊόντα που αναπτύσσουμε τα τελευταία χρόνια, αυτά ποικίλουν από ε, προϊόντα που προέρχονται πολύ γρήγορα, δηλαδή θέσεις πρώτης εντύπωσης. Αυτές συντάσσονται λίγες ώρες μόνο μετά την απεικόνηση, μετά κάποιες άλλες εκθέσεις που χρειαζόμαστε κάποιες μέρες για να τις μετατρέψουμε σε ουσιαστικές πληροφορίες. Και θέλω να πω έτσι χοντρικά ότι περίπου το 40% της δουλειάς μας είναι δεδομένα και το 60% είναι αναλύσεις. Ε, τα δεδομένα δηλαδή και εικόνες δεν είναι και τόσο καθοριστική σημασία για όσους ε, λαμβάνουν αποφάσεις γιατί θέλουν να έχουν αναλυτές που ε, μεταφέρουν αυτές τις φωτογραφίες σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε μια υπηρεσία, προσφέρουμε αυτό τον τεράστιο όγκο πληροφοριών και αυτές τις ε, φωτογραφίες τις ε, αναλύουμε, τις μετατρέπουμε σε πληροφορία χρήσιμη για τον τελικό χρήστη, με και βέβαια και μέσα στο απαραίτητο χρονικό διάστημα. Δεν χρησιμοποιούμε λοιπόν μόνο φωτογραφίες, αλλά χρησιμοποιούμε και αναλύσεις από ε, συνθετικά, γεωγρα... συνθετικά ραντάρ, ε, γεωτερμικές ε, εικόνες, ε, χάρτες, διανύσματα. γενικότερα χρησιμοποιούμε δεδομένα με βάση πάρα πολλές πηγές και καταλήγουμε σε προϊόντα που στέλνουμε στους χρήστες. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα, πολύ πρόσφατο το ένα ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων μας ανέθεσε να στηρίξουμε τους επιθεωρητές στη Συρία που επιθεωρούσαν αποθήκες χημικών όπλων. Ε, και ανέφερε το αίτημα ότι το ε, προϊόν είναι βέβαια ε, μη διαβαθμισμένο, αλλά απευθύνεται μόνο για δημόσια χρήση και έπρεπε εμείς να ανταποκριθούμε γρήγορα. Ε, μπορώ να πω ότι ανταποκριθήκαμε και αυτή τη στιγμή νομίζω γίνεται πολύ σημαντική δουλειά σε επίπεδο Συμβουλίου για την επέκταση αυτής της επιχείρησης ε, μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Σε μια τέτοια περίπτωση κάνουμε το εξής, καθορίζουμε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιθεωρητές και εντοπίζουμε βέβαια τα βασικότερα χαρακτηριστικά, ε, κυρίως ε, στοιχεία ε, που έχουν σχέση με εγκαταστάσεις, αλλά και με άλλα δεδομένα. Μια τέτοια ανάλυση η εμπορική ανάλυση, ε, προφανώς τελική ανάλυση μπορεί να οδηγεί σε μη διαβαθμισμένα έγγραφα και αυτό ε, μας διευκολύνει στο να κάνουμε δουλειά μας ευκολότερα. Αυτό που μπορεί να κάνει ένα δορυφορικό κέντρο, έχει μια ομάδα αναλυτών βέβαια και είμαστε πολύ περήφανοι για αυτούς, μπορούμε να κάνουμε μια συγκριτική ανάλυση μέσα στο χρόνο, δηλαδή πώς ακριβώς έχει αλλάξει μια κατάσταση και νομίζω ότι αυτό βοηθάει επιτόπου τους επιτροπητές να κάνουν και αυτοί καλύτερα τη δουλειά τους όπως το ζητούν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτά τα προϊόντα βέβαια είναι χρήσιμα σε ε, αγροτικές αλλά και σε αστικές περιοχές. Ε, καταλαβαίνετε ότι ε, λόγω του πολέμου στη Συρία είναι σχεδόν αδύνατο να έχει κανείς έτσι μια γενική εικόνα των περιοχών που επιθυμεί να επιθεωρήσει. Γι' αυτό λοιπόν είναι χρήσιμο να υπάρχει υποστήριξη από το διάστημα. Πριν από αυτό, τα Ηνωμένα Έθνη μας ανέθεσαν ε, μία αποστολή. Είχαμε μία τότε την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, πριν από κάποιους μήνες μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε. Τους βοηθήσαμε μέχρι το τέλος, μέχρι να ολοκληρωθεί η ε, αποστολή που αυτή ήταν στη Δαμασκό και μετά έπρεπε να φύγουν. Και η αντίδραση από τους επιθεωρητές είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι επιθεωρητές ε, ε, βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στα προϊόντα, το, τα δορυφορικά προϊόντα. βλέπετε λοιπόν εδώ ε, τις διαφάνειες που δώσαμε για ε, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία εξέπληξαν το προσωπικό των ΗΠΑ ε, που και αυτοί ε, πήγαιναν σε διάφορα μέρη αλλά είχαν στα χέρια τους αναλύσεις για τις εξελίξεις στη χώρα και τα στοιχεία που είχαν τους βοήθησαν επίσης και για να παρλητεύσουν κάποιες δικές τους εικασίες. Άλλα προϊόντα δικά μας είναι τα εξής κάτι που είναι περιζήτητο, κυρίως ε, για όσους ε, βρίσκονται σε αποστολές. Οι χάρτες, εμείς δεν είμαστε κέντρο χαρτογράφησης, όμως είμαστε ένα κέντρο που μπορούμε με βάση τις ε, δορυφορικέ απεικονίσεις να προσφέρουμε βασικούς χάρτες. Επίσης, αυτό που αποκαλούμε borderization, δηλαδή έχει σχέση με τα σύνορα. Όταν τα ε, να ε, ρυθμίσουμε, να τοποθετηθούμε σε θέματα σύνορων, ε, προσφέρουμε και εμείς στοιχεία έτσι ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να έχουν μια αντικειμενική άποψη. Έχουμε και τρισδιάστατα μοντέλα Εδώ λοιπόν βλέπετε ένα παράδειγμα από ένα φράγμα στην Γεωργία που έπρεπε να επισκευαστεί. Οι δύο πλευρές δεν συμφωνούσαν σχετικά με την επισκευή και εμεί τους δείξαμε, κάναμε μία τρισδιάστατη επίδειξη για να ξέρουν τι θα γίνει αν δεν επισκευαστεί αυτό το φράγμα, ε, πώς θα ε, πλημμύριζαν τα χωριά. Βεβαίως οι δορυφορικές απεικονίσεις βοηθούν πάρα πολύ. Εκτός από τις φωτογραφίες χρησιμοποιούμε και άλλα δεδομένα, υπέρυθρες φωτογραφίες. Μερικές φορές αναφέρουμε βέβαια την πηγή, γιατί έτσι μπορεί κανείς να αποκτήσει καλύτερη εικόνα των δραστηριοτήτων. Εδώ έχετε ένα παράδειγμα μια εικόνα SAR ε, που χρησιμοποιείται για την ανάλυση δραστηριοτήτων. Επίσης ε, έχουμε και την δυνατότητα σύγκρισης ε, φωτογραφιών σε διάφορες ημερομηνίε και έτσι μπορούμε να λύσουμε τι εντωμεταξύ έχει διαδραματιστεί να ενημερώσουμε τους αρμόδιους. Οι εικόνες SAR από ραντάρ είναι πολύ δύσκολο να αναλυθούν ε, οι εικόνες ραντάρ συνθετικού ανοίγματο. Και για να είναι βανάγνωστο το αποτέλεσμα, ε, ο αναλυτής ε, χρειάζεται να έχει εκπαιδευτεί 4 μέχρι 6 χρόνια και γενική εκπαίδευση και άλλο ένα χρόνο στα συστήματα SART, συστήματα ραντάρ συνθετικού ανοίγματο. Βλέπετε όμως ότι με τον τρόπο αυτό έχουμε πρώτης κλάσης ε, αναλυτέ ε, στο κέντρο μας. Αυτά που σας λέω τα χρειαζόμαστε εμείς στο κέντρο, αλλά από ό,τι φαίνεται και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν μιλάμε σε συναντέλφους από άλλα κέντρα, όλοι συμφωνούν ότι ενώ υπάρχουν ε, ε, δεδομένα υψηλή ευκρίνειας, ε, υπάρχει έλλειψη αναλυτικών δυνατοτήτων. Σήμερα οι λαμβάνοντες αποφάσεις επιθυμούν να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία και είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν και οι απαραίτητοι πόροι. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι τα νέα προγράμματα σχετικά με το διάστημα και την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, αναφέρομαι και εγώ, συνεχίζω από εκεί που σταματήσαμε για τον Κοπέρνικους, να σας πω ότι το Διαστημικό Κέντρο ε, ασχολείται με εξερευνητικά προγράμματα στην προεπιχειρησιακή φάση. Εμείς ε, παράγουμε προϊόντα τα οποία ε, νομίζω για 7 περίπου χρόνια βρίσκονται στην υπηρεσία του συστήματος ε, Κοπέρνικους. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ασφάλειας και προσβλέπουμε με ανυπομονησία τη συζήτηση ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την τελική μορφή που θα λάβει το Κοπέρνικους. Επίσης θέλω να υπογραμμίσω και ότι η διαχείριση του Κοπέρνικους είναι πολύ σημαντική. <clears throat> να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να στηρίζει μια συγκεκριμένη πολιτική, στην δική μας την περίπτωση ε, την ΚΠΑ, ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προς κλάση προϊόντα που τελικά όμως δεν θα φτάνουν στον τελικό χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος ε, να μην γίνεται η βέλτιστη χρήση αυτού του πολύ καλού προγράμματος. Τέλος, όσον αφορά την ευαισθητοποίηση και την συνειδητοποίηση αναφέραμε ε, ότι το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο <clears throat> πώς πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δουλεύει από πάνω προς τα κάτω, από το διάστημα προς τα κάτω. Κανονικά δουλεύουμε διαφορετικά με τα τηλεσκόπια που στρέφονται προς τα πάνω. Ε, έχουμε όμως εμπειρία σχετικά με τα διαβαθμισμένα και μη διαβαθμισμένα ε, στοιχεία. Ε, προσπαθούμε να τα χρησιμοποιούμε και όσον αφορά τη διαχείριση πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετή εμπειρία. Περιμένουμε και την απόφαση των κρατών μελών για το τι θα γίνει τελικά με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση. Μιλάμε βέβαια και για υποϋπηρεσίες, υπάρχουν αιτήματα για τις υπερπτήσεις δορυφόρων. Αυτό το χρειάζονται πάρα πολύ, κυρίως αυτοί που θέλουν να γνωρίζουν ε, τι συμβαίνει πάνω από, τον, πάνω από μας. Ε, τα χρειάζονται αυτά ε, για να μπορούν να προβλέπουν καταστάσεις σε σχέση με το διάστημα. Ανακεφαλαιώντας κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε μια υπηρεσία του Συμβουλίου με περιορισμένους πόρους, 16,7 εκατομμύρια ευρώ είναι ο ετήσιας ε, ε, προπολογισμό μας. Έχουμε 108 υπαλλήλους. είναι πολύ μετριοπατής ο, ο μα. μας. και προσφέρουμε όλο και περισσότερα ε, γιατί δεχόμεθα όλο και περισσότερα αιτήματα. Ε, θέλουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξη στο μέλλον, ε, θέλουμε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των τελικών χρηστών και να είμαστε σίγουροι ότι η ποιότητα που προσφέρουμε θα βελτιώνεται συνεχώς. Όσον αφορά στη χρήση του διαστήματος, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα έχει επιτύχει θαυμάσια αποτελέσματα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το δρόμο και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη μου χαρά ε, να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις σας. merci, monsieur Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Μερικά μπορεί να σας φανούν ε, λεπτομέρειες από αυτά θα πω, αλλά θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μπρουνέ πρώτα απ' όλα να μου πει κατά πόσο το πλαίσιο, η πρόσφατη επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει, με το περίφημο σκάνδαλο για την Ενέσα. Αυτού του είδους οι πληροφορίες που δείχνουν πόσο ευάλωτα είναι τα κράτη-μέλη για κάτι που δεν έχει απόλυτα σχέση βέβαια με τη δορυφορική δραστηριότητα, αλλά έχει να κάνει με τα δεδομένα γενικά, θα μπορούσε να ήταν και δορυφορικά. Αυτό το πλαίσιο πιστεύετε ότι μπορεί να ευνοήσει τη συνδυτοποίηση των χωρών μελών για τη σημασία που έχουν τέτοια προγράμματα και να κάνει τα κράτη-μέλη να παίξουν καλύτερα το παιχνίδι, είτε πρόκειται για τη χρηματοδότηση, είτε πρόκειται για την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσει περισσότερο προς τέτοιου είδου προγράμματα. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Επίσης, αναφερθήκατε στη Eurosur. Κόνοψ. Θέλω να σας ρωτήσω όσον αφορά την αλυσίδα εντολών και τη συλλογή πληροφοριών. Ίσως ο κύριος Λοβέντσιτς να έχει να μας πει επίσης περισσότερα. Πώς γίνεται η οργάνωση, πώς συλλέγονται καταρχήν τα δορυφορικά δεδομένα, υποθέτω μέσω απεικόνησης, σε ποιο καλάθι πέφτουν, ποιος τα παίρνει, πώς κυκλοφορεί η πληροφορία και πού φτάνει. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι αυτή τη διαδρομή. Μπορείτε. Και κάτι άλλο που σκέφτηκα. Σε σχέση με τις διάφορες επιχειρήσεις, τους χώρους επιχειρήσεων. Σήμερα έχουμε ένα πρόβλημα με μια περίπτωση, όπου είμαστε περίπου τυφλοί, ενώ ακριβώς θα θέλαμε να μπορούμε να βλέπουμε πιο καθαρά. Πρόκειται για τη Λιβύη. Είχαμε μια αποστολή, ΚΠΑ, που δυσκολεύτηκε να αναπτυχθεί ακριβώς επειδή υπάρχει αστάθεια στη Λιβύη σήμερα και θεσμικά δεν έχουμε συνομιλητή εκεί. Η αποστολή όμως που έχει ως στόχο να ελέγξει καλύτερα τα σύνορα της Λιβύης μας φέρνει αντιμέτωπος με τεράστιες προκλήσεις, τα νότια σύνορα της Λιβύης Δηλαδή, μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε άπαξ και αναπτυχθεί, ακόμα και αν δεν λειτουργήσει πλήρως η αποστολή, μπορεί να στηριχτεί στο ΣΑΤΣΕΝΤ για να ξεκινήσει τις εκτιμήσεις, την αξιολόγηση και να μπορέσει να λειτουργήσει, ακόμα βέβαια και αν οι συνθήκες ανάπτυξης αποστολής είναι πολύ δύσκολες. Και τελευταία μου ερώτηση. Αναφερθήκατε σε διάφορες πηγές για το ΣΑΤΣΕΝΤ. Πιστεύετε ότι κάποια μέρα θα μπορούσαμε να δούμε τα κράτη, ίσως όχι από κοινού, αλλά τουλάχιστον να μπορούν να σας δώσουν ε, βάση μη επανδρομένων ε, ε, σκαφών στοιχεία για την εποπτεία των ζωνών όπου έχουμε επιχειρήσεις. Είναι κάτι το οποίο τίθεται σαν υπόθεση. Μπορεί να υπάρξει κάποια μέρα αυτό στο μέλλον. Και δευτερευόντως, άλλη μια ερώτηση. Αυτή είναι μια δυνατότητα που μπορούμε να φανταστούμε και εκτιμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί οι επιτροποί αναφέρθηκαν. Πολλές φορές είπαν ότι δεν θα ήταν άχρηστο να έχουμε τέτοια μη επανδρομένα σκάφη ως Ευρωπαϊκή Ένωση για την εποπτεία μη στρατιωτικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν το ΣΑΤΣΕΝ θα μπορούσε να αποτελέσει έναν παράγοντα λειτουργίας. Κύριε Τσέμκε, έχετε ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα καταρχήν να, να ευχαριστήσω θερμά τους καλεσμένους μας για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας έδωσαν και να κάνω μια ερώτηση κάπως ε, διαφορετικού χαρακτήρα. Οι περιπτώσεις του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικους ε, μας δείχνει ότι βρισκόμαστε ακόμη σε φάση δημιουργίας των δύο συστημάτων. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό εδώ είναι ο χρόνος και ο ρυθμός δημιουργίας αυτών των συστημάτων. Μιλούμε για τεχνικές πολύ εξεζητημένες, πολύ προηγμένες. Οπότε μερικές φορές η καθυστέρηση, η μεγάλη παράταση δημιουργεί πρόβλημα γιατί στα συστήματα αυτά έχουμε στοιχεία με διαφορετικές ε, τεχνικές ικανότητες. Σχετικά πρόσφατα εγκρίναμε τον κανονισμό, ε, εγκρίναμε μάλλον τον προϋπολογισμό για το 2014-2020, το πολιτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε γνωρίζουμε ήδη σήμερα ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχω ερώτηση προς τον δόκτωρα Μπρουνέτ. Έχετε πια για τον από τον προϋπολογισμό συγκεκριμένα κονδύλια για τα δύο συστήματα. Με τα κονδύλια αυτά, τι μπορείτε να πραγματοποιήσετε για το Γαλιλαίο και τον Κοπέρνικος και τι δεν θα χρηματοδοτηθεί εξαιτίας έλλειψης πόρων. Merci. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπλουνέ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Τανζό. Πρώτον, ο παραλληλισμός που κάνατε. Με την ΕΝΕΣΑ. Οι δορυφόροι βέβαια πιάνουν διάφορες ε, επικοινωνίες δορυφορικές και προβληματική συστημάτων όπως είναι ο Γαλιλαίος, ο Κοπέρνικος ή το SST, μπορεί να έχουν διαφορές αλλά έχουν και πολλά κοινά. Στην περίπτωση της NSA συνδυτοποίησαμε ή νομίζαμε ότι συνειδητοποίησαμε ότι κάναμε πάντα, ότι κάναμε και κατά το παρελθόν αλλά με τεχνολογικά μέσα που δεν φανταζόμασταν και με δυνατότητες φοβερές σε σχέση με το παρελθόν. Οπότε, το πρώτο που συνειδητοποίησαμε σε αυτό που συζητάμε και κυρίως για το SST, εποπτείες δηλαδή και χνηλάτησης, είναι ότι αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Θέλουμε να φτάσουμε σε δυνατότητες συγκρίσιμες με αυτές που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εφόσον η ερώτηση λοιπόν είναι αυτή, η απάντηση είναι όχι. Δεν θα είμαστε σε θέση. Δεύτερον, πρόσβαση στα δεδομένα. Όπως είδαμε όλα αυτά τα συστήματα προσφέρουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων που αρχαιοθετούνται, επεξεργάζονται και πρέπει να είναι διαθέσιμα την κατάλληλη στιγμή για τον κατάλληλο άνθρωπο. Σήμερα λοιπόν στα διάφορα συστήματα, και αυτό είναι και το πρόβλημα του συστήματος επαπίας και, και δείχνει η απάντηση λοιπόν και εδώ είναι πως όχι. Για να γίνει και πάλι ο παραλυσμός αυτός, μπορεί να είναι βέβαια πιο πολιτικό το ζήτημα, αλλά αυτό είναι για την υπηρεσία εξωτερική δράση. Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανεί στη συνεργασία, στη μη συνεργασία με τους, διεθνούς μα με τους διεθνείς μας εταίρους. Αυτό όμω που για μένα είναι προφανές είναι ότι το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες, στην τεχνολογική ανάπτυξη, και όλα έχουν να κάνουν με την αρχιοθέτηση και την υπερσυρασία των δεδομένων έχουν σαν αποτέλεσμα τα συστήματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίος και ιδιαίτερα στο SST αν δεν υπάρχει συντονισμός και κοινοτικοποίηση κατά κάποιο τρόπο του Κοπέρνικου δηλαδή και του Γαλιλαίου ποτέ δεν θα φτάσουμε να έχουμε κάτι αντίστοιχο. Τώρα έρχομαι στη δικιά σας ερώτηση για την υπηρεσία ασφάλειας κυρίως και για τη Eurosur. Αυτό που εμείς κάνουμε επί του παρόντος είναι ότι αφού ήρθαμε σε επαφή με τους ενδυνάμει χρήστες, τους υποψήφιους χρήστες, προχωρήσαμε σε τεχνικές συστάσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν όχι μόνο με τον τύπο των δεδομένων που θέλουμε να έχουμε, αλλά και με, το, με ποιον τρόπο θα επεξεργαστούμε και ποιος θα επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά. Οπότε εδώ ο φυσικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να είναι η Frontex. Συνεπώς μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε ότι όπως έγινε και με το Γαλιλαίο ή με την κρατικά υπηρεσία θα υπάρξουν κάποιοι εταίροι που θα έχουν πρόσβαση και η Frontex μπορεί κατά προτεραιότητα ή και αποκλειστικά να έχει στη διάθεσή της κάποια δεδομένα. Σήμερα πάντως από τις έξι του Κοπέρνικου, εκείνη για τα κατεπήγοντα ή για την δαφική επικράτεια που λειτουργούν, είναι ένα θέμα, ενώ για την ασφάλεια θα πρέπει να αναπτύξουμε βάση τεχνικών συστάσεων που έχουν εισαχθεί, θα δούμε στη συνέχεια πώς θα προχωρήσουμε, πώς δηλαδή το σύνολο των δεδομένων θα πηγαίνει στη Frontex και πώς θα τυχαίνει επεξεργασία. Έρχομαι τώρα στην χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών. Έχετε δίκιο γιατί φτάνοντας εκεί που βρίσκομαι τώρα, σε αυτή τη θέση δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να βάλουμε από κοινού, όχι δεν πρόκειται για συγχώνευση, αλλά πρόκειται για μια εναρμονισμένη ανάπτυξη κύκλων που δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Ο δημοσιονομικός ευρωπαϊκός κύκλος, για παράδειγμα, που είναι τήσιος ή εφταετής και ο κύκλος τεχνολογικής ανάπτυξης που περιλαμβάνει και την διαστημική έρευνα έχει ως αποτέλεσμα Έχουμε το μακροπρόθεσμο σενάριο με το οποίο λίγο πολύ ζητάμε από την Επιτροπή να δεσμευτεί για δαπάνες που ίσως προβλεφθούν στα μέσα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Όχι αυτόν που έρχεται, το επόμενο. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο καθένας, η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να βλέπουν τον Κοπένικο και τον Γαλιλαίο και σαν βιομηχανικό πρόγραμμα, αλλά και σε κάτι που για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία νίκη ο Γαλιλαίος και που μεθαύριο μπορεί να γίνει και ιδιοκτήτρια ή να νοικιάσει τέλο πάντων δορυφόρους ε, Κοπέρνικου, θα γίνει πάροχος υπηρεσιών. Οπότε το μόνο που χρειάζεται είναι να διασφαλίσει τη συνέχεια της υπηρεσίας αυτής και την ε, διάρκεια ζωής. Συνεπώς πρέπει μαζί να μπορέσουμε να δώσουμε εγγυήσει. Δεν λέω να αλλάξει ο δημοσιονομικός κανονισμός ή κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αναλάβουμε πολιτικές δεσμεύσεις ώστε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια αυτή της υπηρεσίας που θα προσφέρουμε. Ο αντιπρόεδρος Γιάννη το είπε αρκετές φορές ότι περιμένουμε πολλά από την ε, ανάπτυξη την θαλάσσια του Κοπέρνικου και σε θέματα άμυνας και σε θέματα μη στρατιωτικά. Δεν μπορούμε πάντως να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις να επενδύσουν για βάση δεδομένων που θα τους προσφέρουμε και μετά να πούμε ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να τους δίνουμε τα δεδομένα τα οποία θέλουν. Εκεί θα υπήρχε πρόβλημα. Πιο συγκεκριμένα, Σήμερα έχουμε τις αρχικές ε, ε, επιχειρήσεις, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για παράδειγμα και έχουμε το σύνολο των δορυφόρων και τις περισσότερες ε, νέες εκδοξεύσεις που έχουν πληρωθεί μέχρι τα μέσα του επόμενου οικονομικού κύκλου. Βάσει λοιπόν του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου που αρχίζει τον Ιανουάριο, θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη χρηματοδότηση δορυφόρων που έχουν ήδη προβλεφθεί για την επόμενη επταετία. Είναι προφανές ότι τότε, στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, η ζωή ενός δορυφόρου είναι γνωστή. 7 με 10 χρόνια είναι η διάρκεια ζωής του. Στο μεταξύ λοιπόν πρέπει να βρούμε την πολιτική δέσμευση ώστε να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε τον επόμενο δορυφορικό κύκλο. Και όπως σας είπα στην αρχή υπάρχουν έξι οικογένειες δορυφόρων, οπότε για τέσσερις από αυτές στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου 14 με 20 μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τις δύο ή μάλλον τις τρεις πρώτες μονάδες. Έχουμε δηλαδή κάποιο περιθώριο λιγμών και σας ευχαριστώ που το ρωτήσατε αυτό, γιατί είναι πράγματι πρόβλημα. Πώς θα συνεχίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο προβλέπεται να διαρκεί 15 χρόνια, με ένα προπολογισμό ο οποίο ανανεώνεται ετησίως ή και τόσο πάνω καταρτίζεται ένα γενικό του πλαίσιο κάθε 7 χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το κέντρο δορυφόρων είναι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους και πολύ δραστήριο στην εξασφάλιση της προστασίας των συστημάτων ασφαλείας. Και αυτά εφαρμόζονται πλήρως στο δορυφορικό κέντρο. Οπότε η εμπιστευτικότητα, κεραιότητα, προσπελασιμότητα είναι βασικοί στόχοι που εκπληρώνονται. Επιπλέον, τα ασφαλή δίκτυα που επιτρέπουν ε, ε, τη μεταφορά διαβαθμισμένων δεδομένων στις ε, διαφερόμενους συγκεντρώνει λίγους φορείς, κυρίως επιχειρησιακά κέντρα και αρχηγεία, αλλά δεν συνδέει πρωτεύουσες στα κράτη-μέλη. Οπότε είναι ύψητη προτεραιότητα η επέκταση αυτού του συστήματος και στις πρωτεύουσε. και η ανάπτυξή του ανάλογα με το βαθμό των απαιτήσεων και των αναγκών των κρατών μελών και τη συνεργασία τους με τα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Όλα τα στοιχεία ενός συστήματος ασφάλειας θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως, όχι μόνο το τμήμα πληροφοριών και επικοινωνιών, αλλά το σύστημα ολόκληρο, το θέμα της ηλικής ασφάλειας είναι σημαντικό. Και υπάρχουν όλο και αυξανόμενες ανάγκες. Και οι συγκεκριμένες επιπτώσεις ε, μη της ασφάλειας είναι η απειλή των επιχειρήσεων και των δράσεων που παρεμπορίζονται από έλλειψη ασφάλειας και πιθανές ζημίες που θα έχουμε στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό είναι η πιστή προτεραιότητα αυτή η ασφάλεια. Τώρα, για το ΕΡΟΣΟΥΡ και τη Λιβύη, τη συγκεκριμένη ερώτηση που θέσατε. Θέλουμε συμβουλευτικό χαρακτήρα του οργανισμού που δεν αποφασίζει από ποιους τομείς και από ποιες περιοχές θα συγκεντρώσει τις ε, φωτογραφίες και θα τις αναλύσει. Αυτό είναι μια πολιτική διαδικασία και αφορά την, είπατε, εκπρόσωπο. Εμείς θα εφαρμόσουμε τις πολιτικές αποφάσεις. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τη συνοριοποίηση που σας ανέφερα ή τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σε παράκτιες ζώνες, εκεί επιτύχαμε σημαντικά πράγματα. Και ήταν σημαντικό το έργο που κάναμε για την Αταλάντη, για την επιχείρηση Αταλάντη και το κέντρο επιχειρήσεων των Northwood. Οπότε έχουμε δημιουργήσει μια μεθοδολογία που μπορεί να εφαρμοστεί και στην περίπτωση αυτή και ο συνδυασμό των δεδομένων από πηγές διαστημικές και της συνεργασίας επιτόπου είναι πολύ σημαντική. Τώρα, κανένας δεν θέλει το Κοπέρνικος και το Εροσούρ να είναι μόνο ένα εξαιρετικό επιστημονικό σχέδιο. Εμείς θέλουμε να μην είναι μόνο ένα επιστημονικό σχέδιο, αλλά και ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Και μια, επιχειρη... μια υπηρεσία που θα βελτιώνει την ποιότητα των επιχειρήσεων. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ακούμε τη γνώμη και το feedback από τους τελικούς χρήστες. Αυτό εφαρμόζουμε και στο SatSend. Γιατί πρώτα ακούμε αυτά που μας λένε και μόνο τέτοιες αποστολές αναλαμβάνουμε όταν μας τις αναθέτουν. Ακούμε συγκεκριμένα τους τελικούς χρήστες, τις ανάγκες που έχουμε και αυτές προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε. Και φαντάζομαι και το αεροσούρ αυτό θα κάνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρήση της απεικόνησης ή βίντεων εικόνων από τα μη παδρομένα αεροσκάφη, τα drones. Ήδη υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά μέχρι στιγμής στο κέντρο δορυφόρων, από το κέντρο δορυφόρων δεν ζητήθηκε η ανάλυση τέτοιων ε, βίντεο. Και από νομική άποψη θα πρέπει να εξεταστεί αυτό το θέμα και να λάβουν την απόφαση περιπτωσιολογικά τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, αν ενδιαφέρονται για κοινή διαχείριση των δεδομένων ή να ζητήσουν από το SAT Center τα αναλύσει. Η ανάλυση από μόνη της είναι τεχνικώς εφικτή. Το θέμα είναι αν η διαδικασία λήψη αποφάσεων ή δράσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια ταχεία ροή αναλυμένων, επεξεργασμένων πληροφοριών. Γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει η δρασεων μπορει να χρησιμοποιησει τετοια ταχεια ροη αναλυμενων εξεργασμένων πληροφοριων γιατι κατι τετοιο προυποθετει η ικανοτητα 24 ώρες, 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επίσης, να αναφερθώ σε κάτι που είπατε στην εισαγωγή σας. Υπάρχουν σημαντικά θέματα στην διαστημική μας πολιτική για τα οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι και είναι πρώτης τάξεως διεθνώς. Αλλά αυτή την ε, τεχνολογία, την ευρωπαϊκή τεχνολογία πρώτης τάξης που έχουμε θα πρέπει να την εφαρμόσουμε στι ευρωπαϊκές δράσεις γιατί εκεί είναι που υπάρχει έλλειμμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και οι νομοθετικέ διαδικασίε που αναφέρθηκαν είναι πολύ σημαντικέ ώστε να βελτιώσουμε τη διακυβέρνηση και να αναβαθμίσουμε την αποτελεσματικότητα τη δράση ώστε να φτάσει στο επίπεδο τη προηγμένη τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τηρήσαμε πλήρως το χρονοδιάγραμμα και πιστά. Σας ευχαριστώ θερμά και ήταν πολύ σημαντικό το στατιστικό στοιχείο που μας δώσετε κύριε Λαβρέντζιτς για την, το αυξανόμενο αριθμό των στοιχείων που συγκεντρώνουμε αυτόνομα, γιατί μας ενδιαφέρει η στρατηγική αυτονομία. Είναι μία έννοια που προκαλείται το γέλοτα είτε τον κλαθμό, αλλά είναι σημαντικό αυτό το θέμα της αυτονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μάλιστα μερικοί συνάδελφοι εκπλήσονται με τέτοιου είδους υψηλές, ε, όπως θεωρούν, ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Αλλά γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ και νομίζω ότι και τα δικά σας ε, θεσμικά όργανα και δικοί οργανισμοί αυτό προσπαθούν να κάνουν, να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν και να διατηρήσουν μια τέτοια αυτονομία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος και ταυτόχρονα εξεπλάγει από την ε, εξέλιξη αυτών των στοιχείων. Στην αρχή είχαμε ένα μικρό ποσοστό και έχουμε φτάσει σε 60% των δεδομένων που συγκεντρώνουμε αυτόνομα μόνοι μας. Βέβαια, έχουμε δημοσιονομικά προβλήματα, κάποιες ελλείψεις εκεί. Το μήνυμα ελήφθη και θα ανταποκριθούμε στην έκκλησή σας για να διεκπαιρεώσουμε το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία αυτή, γιατί θα είναι κρίμα να μπλοκαριστούν λόγω καθυστέρησης τόσο στρατηγικής σημασίας προγράμματα. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας και τη συμβολή σας και φαντάζομαι ότι μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε και να εξετάσουμε το σύνολο του τρίτου καλαθιού και ολόκληρο το θέμα του διαστήματος και της πολιτικής που ακολουθούμε μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσουμε μια συνέχεια, να συνεχίσουμε τη συζήτηση και το θέμα το βιομηχανικό είναι σίγουρα το περισσότερο υποσχόμενο θέμα. Θα πρέπει να είμαστε Συγκριτημένα αισιόδοξη για το θέμα το επιχειρησιακό και των ικανοτήτων, αλλά το θέμα το βιομηχανικό είναι σίγουρα πιο προσιτό. Σας ευχαριστώ και σας ανανεώνουμε την πρόσκληση για μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε θερμά πάντως. Δύο δίλεπτη διακοπή για να αποχαιρετήσουμε τους καλεσμένους μας και συνεχίζουμε με το εμπόριο των όπλων. Bien, mesdames, messieurs, nous allons euh, reprendre et terminer. Ερχόμαστε και πάλι στη δουλειά μας. Καθίστε να συνεχίσουμε. Είμαστε τώρα στην συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Ξέρετε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο απασχολεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και αρκετό καιρό. Οι εξελίξεις ήταν ευτυχείς. Με την υπογραφή τελικά της συνθήκης αυτή στα Ηνωμένα Έθνη. Βέβαια δεν υπέγραψαν όλες οι χώρες. Κάποιες προμηθευτές όπλων δεν συμφώνησαν, αλλά ναι. 154 χώρες τελικά τάχθηκαν υπέρ και χρειάζονται 50 επικυρώσεις για να αρχίσει να ισχύει η συνθήκη. Σε είπα ότι το Κοινοβούλιο μας εδώ και χρόνια έχει κινητοποιηθεί για να υπογραφεί αυτή η συνθήκη. Φυσικά και είναι ενδιαφέρον και χαιρετίζουμε το αποτέλεσμα Γι' αυτό και η Υποπιτροπή μα έχει αναλάβει ένα ψήφισμα για το θέμα. Έχουμε και γνωμοδότηση, επίσης όσον αφορά την επικύρωση της συνθήκης. Η Ίντα είναι αρμόδια και ο συνάδελφος Λίζεκ έχει την γνωμοδότηση. Εγώ έχω το πολιτικό ψήφισμα. Το επόμενο θέμα θα το δούμε αμέσως μετά την επικύρωση δηλαδή. Λοιπόν, εμείς εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την υπογραφή, αλλά υπογραμμίζουμε και κάποιες ελλείψεις σε σχέση με τα όσα το κοινοβούλιο μας έχει διεκδικήσει κατά το παρελθόν και όχι μόνο και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία δεν διευκρινίζονται παρκώς όσον αφορά τους ορισμούς. Για πιο πρόκειται δηλαδή ακριβώ κάποιε κατηγορίε όπλων δεν καλύπτονται αρκετά αποτελεσματικά κατά τη γνώμη μα. Θα θέλαμε μια βελτίωση του κειμένου, αλλά βέβαια πολιτικά φυσικά και εκφράζουμε την ικανοποίησή μα για την υπογραφή τη συνθήκη. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά σήμερα. Ο συνάδελφος Λίζικ δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Υπενθυμίζω και πάλι ότι η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου έχει αναλάβει την διαδικασία επικύρωσης της συνθήκης για το εμπόριο όπλων, μια που πρόκειται για διεθνές εμπόριο, έτσι. Για την επικύρωση εμείς γνωμοδοτούμε μόνο. Κάτι που έχει αναλάβει ο κύριος Λίζεκ. Το βασικό της συνθήκης είναι ότι τα σεβαλόμενα μέρη πρέπει να έχουν ένα εθνικό σύστημα ελέγχου των συμβατικών όπλων που αξιολογούν πριν δοθεί άδεια. Αξιολογούν δηλαδή τον κίνδυνο από τα όπλα αυτά στην ειρήνη και την ασφάλεια την περίπτωση να ε, οδηγήσουν σε σημαντική παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τρομοκρατικών ε, ενεργειών ή εγκληματικών ε, ενεργειών που εμπίπτουν στο διεθνές έγκλημα. Η γνωμοδότησή μας δεν μπορεί παρά να είναι θετική βέβαια. Αυτά μου ζήτησε ο κύριος Λίζεκ να σας πω. Φαντάζομαι δεν έχετε αντίρρηση για το περιεχόμενο της γνωμοδότησης. Έτσι κι αλλιώς πάντα οι απόντες έχουν άδικο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιαναμάκη, η οποία συνέταξε το 2012 ένα ψήφισμα που είχε να κάνει με τις διατάξεις αυτές του κειμένου της συνθήκης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Λίζεκα που απουσιάζει. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο για το ψήφισμα και τη γνωμοδότηση που συντάξατε. Εγώ Είμαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και χωρίς πρόβλημα θα συμφωνήσω με τις ιδέες που παραθέτει ο Πρόεδρος στη γνωμοδότησή του. Χαιρόμαστε που η συνθήκη για το εμπόριο των όπλων επιτέλους και μετά από αρκετές δυσκολίες έχει συναυθεί Οπότε λαμβάνονται υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Κάτι άλλο θετικό είναι ότι η συνθήκη περιλαμβάνει υποχρέωση εκτενούς ενημέρωσης για τις διάφορες πρακτικές. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μία συνθήκη ε, δεν θα είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης υποβολής εκθέσεων. Τώρα θα πρέπει να επενδύσουμε και στο θέμα της παρατήρησης. Ε, δηλαδή να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή της συνθήκης. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μεριμνήσει ώστε και τα κράτη-μέλη της ε, να δώσουν το καλό παράδειγμα της εφαρμογής αυτής της συνθήκης. Και χαίρομαι που τα πυρομαχικά και τα εξαρτήματα των όπλων συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη γιατί έχουν αντίστοιχο ρόλο με αυτό των όπλων. Βέβαια είναι αρνητικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συνθήκη. Η συνθήκη θα ήταν πιο ολοκληρωμένη αν την προσυπόγραφαν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι περιφερειακοί εταίροι μας. Ήδη αρκετές χώρες έχουν υπογράψει τη συνθήκη. Θα πρέπει τώρα να, να περάσουμε στη διαδικασία της κύρωσης. Φαντάζομαι ότι όσοι υπέγραψαν τη συνθήκη θα την κυρώσουν και μετά θα περάσουμε στη φάση της εφαρμογής. Ελπίζω να υλοποιηθεί και αυτή η φάση της έμπρακτης εφαρμογής και να μην παραμείνει μια συνθήκη στα χαρτιά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρκετέ ε, χώρε μέλη που φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερω για την εφαρμογή τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστώ ότι μετά την υπογραφή και την κύρωση τη συνθήκη θα ισχύσουν στην πράξη και οι κανόνε τη και θα τηρηθούν οι λιμένε δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Ευχαριστώ θερμά και τον Πρόεδρο, παραλαμβάνω, για τη γνωμοδότησή του. Σας ευχαριστούμε κυρία Γετενμάκη. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Γκάρσλαντ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, αν δεν κάνω λάθο, εσείς παρακολουθείτε αυτή την υπόθεση, αυτό το θέμα. Σα ευχαριστώ. Η έγκριση της συνθήκης αυτής τον Βίλιο μετά από 7 χρόνια συζητήσεις και διαπραγματεύσεις στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση που να ξέρετε ότι στήριξε τη διαδικασία καθόλου την πορεία. Με δραστηριότητες από τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου υπέρ της στήριξης της συνθήκης για το εμπόριο όπλων με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι δραστηριότητες αυτές βέβαια βοήθησαν στη συνδυτοποίηση για τη διαδικασία της συνθήκη αυτής για να διευρυνθεί και ε, το, οι χώρες οι οποίες στηρίζουν τη συνθήκη αυτή. Επίσης για να ισχυθεί η διαφάνεια και να υπάρξει και η προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε ενεργά στις πέντε προπασκευαστικές επιτροπές από το 2009 μέχρι το 2012 και στην ε, τελευταία ε, διάσκεψη το Μάρτιο του 2013. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ε, είτε συντονισμός με τις χώρες μέλη, είτε το κεκτημένο των ελέγχων που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεκτημένο αυτό έχει να κάνει με την κοινή θέση για το εμπόριο όπλων με τρίτες χώρες αλλά υπάρχει και η 2009 του 43 όσον αφορά το εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού. Η συνθήκη που τελικά ε, συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένα ισορροπημένο και εύρωστο εργαλείο. Και είναι εύρωστο γιατί περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια όσον αφορά το διεθνή ανθρωπιστικό δίκαιο και περιλαμβάνει απαγορεύσεις για μεταφορές που θα παραβίαζαν τον διεθνή ανθρωπιστικό δίκαιο. Πολλά καλύπτονται από τη συνθήκη, περιλαμβάνονται και τα πυρομαχικά και τα συστατικά των όπλων. Επίσης περιλαμβάνεται το θέμα της διαφάνειας η συνθήκη αυτή μπορεί να λειτουργήσει γιατί συνάδει με τα όσα αναφέρει και το κοινοτικό δίκαιο, για παράδειγμα για ε, τα όπλα. Είναι επίσης η συνθήκη αυτή ανοιχτή, μάλλον δεν πετύχαμε να ανοιχτεί και σε άλλους οργανισμούς, κυρίως γιατί η Κίνα αντιτάχθηκε σε αυτό. Αν πάντως θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε πρέπει να έχουμε την υπόψη μας, να υπόψη ότι έξι χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ μπορεί να τροποποιηθεί η συνθήκη αυτή. Κάτι ε, το οποίο θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεληθεί όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλες ομάδες όπως είναι η Καραϊβική ή οι χώρες της Δυτικής Αφρικής. Νωρίτερα αναφέρθηκα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Είναι σαφές ότι οι προδιαγραφέ τη συνθήκη αυτή είναι χαμηλότερες από αυτές που σχίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το εύρο εφαρμογή κλπ. Αλλά η συνθήκη όμως για πρώτη φορά βάζει κοινέ διεθνεί προδιαγραφές και θέτει ένα πλαίσιο για να συζητιόνται θέματα που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής η αξιολόγηση μέχρι τώρα λέει ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνάδει απόλυτα με τη συνθήκη αυτή, εμπορίας όπλων, λαμβάνοντας υπόψη τόσα περιλαμβάνει η συνθήκη που λέει ότι πρέπει να παραμείνουν τα εθνικά συστήματα. Είναι σημαντικό να θυμηθούμε εδώ ότι η συνθήκη για το εμπόριο όπλων είναι μια βάση, δεν είναι μια οροφή. Αν επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές χρειάζονται για να δούμε πώς θα εφαρμοστούν συγκεκριμένα τα κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου που προβλέπει η συνθήκη. Η αξιολόγησή μας μέχρι τώρα λέει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε επίπεδο εγχειριδίου Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνουν το τι ισχύει σε εθνικό επίπεδο. Μια τέτοια αξιολόγηση συμβατότητας είναι πολύ σημαντική, μια που χρειάζεται η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην απόφαση του Συμβουλίου να επιτρέψει τα κράτη-μέλη να επικυρώσουν. Οι χώρες ε, μέλη έχουν όλες κυρώσει τη συνθήκη και είναι πολύ σημαντικό που ήμασταν από τους πρώτους. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, επιθυμούν να τεθεί γρήγορα σε αυτή η συμφωνία, διότι οι αρχικές αποφάσεις ε, θα ληφθούν από τις πρώτες ε, από τις χώρες που θα ε, υπογράψουν αυτή τη συνθήκη. Ας έρθω τώρα στην ευρύτερη προοπτική εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σαφές ότι η συνθήκη αυτή υποστηρίζεται διεθνώς και μέχρι σήμερα έχουμε 115 κράτη που έχουν υπογράψει και 8 έχουν επικυρώσει και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό ως αποτέλεσμα γιατί δεν έχουν περάσει ούτε 6 μήνες από τις πρώτες υπογραφές. Βέβαια, ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και προβλήματα. Και εδώ παραθέτω αυτά που είπε μία ΜΚΟ στην, υπογραφή, στην τελετή υπογραφή 3 Ιουνίου που είπαν ότι ε, η υπογραφή αυτή της συνθήκης δεν σημαίνει ότι σταματάει το εμπόριο, απλά η αρχή του τέλους. Και υπάρχουν τρία τέτοια προβλήματα. Πρώτον, ε, ότι υπάρχουν τα εύκολα προβλήματα, δηλαδή να τεθεί η συνθήκη σε ισχύ, άρα δηλαδή οι 50 που υπολείπονται να επικυρώσουν το στομότερο δυνατόν. Υπάρχει κάποια κινητικότητα σε διεθνές επίπεδο και αναμένεται και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα μέχρι το τέλος του 2014 θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη. Δύο άλλα προβλήματα είναι η υποστήριξη και η ε, σωστή εφαρμογή και η διάδοση της συνθήκης. Ε, η αποτελεσματική εφαρμογή απαιτεί τα κράτη να μπορούν να ελέγχουν ελέγχουν τη ροή των όπλων από και προς την επικράτειά τους. Επίσης αυτά έχουν επιπτώσεις και είναι σαφές ότι ένας μεγάλος αριθμός κρατών χρειάζονται σημαντικές, σε σημαντική νομική και ε, διοικητική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν τη συνθήκη αποτελεσματικά. Η διάδοση της συνθήκης έχει σημασία, διότι το να ρυθμίζει κανείς το εμπόριο των όπλων, αυτό είναι εξορισμού ε, ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν η συμβολή της ε, συνθήκης ε, δεν σημαίνει κάτι το απόλυτο και αυτό που έχει σημασία είναι να περιλαμβάνονται, να ρυθμίζονται τα θέματα των σημαντικών εμπόρων. Ξέρετε χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία τον Απρίλιο του 2013 δήλωσαν ε, αποχή στην ψηφοφορία και αυτό ε, δημιουργεί προβλήματα ε, ως προς την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η συνθήκη αφορά και εξετάζει όλες τις διπλωματικές δυνατότητες και τις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες έχουν κατατεθεί διαβήματα το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει βέβαια τώρα τύχη επεξεργασία και πρόκειται να υποβληθεί στο Συμβούλιο. Θα υποστηρίζει κρατή που επιθυμούν να έχουν αυστηρότερα συστήματα μεταφοράς όπλων με στόχο ε, να γίνεται και σωστή εφαρμογή της συνθήκης. Οι προσπάθειες αυτές ε, και τα αποτελέσματα θα εξεταστούν σε ένα ευρύτερο περιφερειακό και θεσμικό πλαίσιο όπου θα συγκεντρωθούν χώρες, κυρίως αυτές που είναι επιφυλακτικές απέναντι στη συνθήκη για να μπορεί να ασκηθεί πίεση από τους ομότιμους τους. Και παράλληλα με αυτές τις δραστηριότητες που πρέπει να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα, άμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει κυρίως όταν τα κράτη-μέλη θα κατεθέσουν την επικύρωση και έτσι θα υπάρχουν περισσότερε δυνατότητε θέση, σε ισχύ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Η υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών στη συνθήκη είναι ένα κοινό εγχείρημα από κοινού με άλλε χώρε. Από τι πρώτε ή από τι 115 που υπέγραψαν, πάνω από 30 είναι Αφρικανικέ, 20 Λατινική Αμερική και καραϊβική. Αυτέ έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα λόγω τη του εμπορίου. Η δέσμευση προς τη συνθήκη καταδεικνύει ότι η διεθνή κοινότητα μπορεί να διεκδικήσει ε, την ε, πλήρη, τον πλήρη έλεγχο μέσω της συνθήκη. και έτσι η συνθήκη μπορεί να συμβάλλει ε, στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε διεθνέ επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τον κύριο Μωρό από το Κέντρο Έρευνας για την Έρευνα και την Ασφάλεια στις Βρυξέλλες που παρακολουθεί όλος ιδιαίτερο το θέμα αυτό του εμπόριου των όπλων. Θέλετε μήπως να μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Κυρίε και κύριοι, η διαπραγμάτευση και έγκριση τη συνθήκη για το εμπόριο όπλων είναι το πρώτο βήμα μια μεγάλη διαδικασία προκειμένου να μπορεί να επηρεάσει θετικά τις συνθήκες ζωής και την ασφάλεια του πληθυσμού. Η διαδικασία επικύρωσης βέβαια λαμβάνει χώρα σε πολλές χώρες τώρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα περιμένουμε να αρχίσει να ισχύει. Προς το παρόν όμως πρέπει να τη δούμε αυτή την συνθήκη λαμβάνοντας υπόψη και τις αδυναμίες της, αλλά και τις δυνατότητες ερμηνείας που παραμένουν ανεκτές. Επίσης παραμένουν προκλήσεις με τις οποίες θα έρθουν αντιμέτωποι αντιμέτωπα τα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι ένα κείμενο ατελές, το οποίο αποτελεί τον συμβασμό μεταξύ 190 χωρών. Το κείμενο περιλαμβάνει πρόοδο βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο του εμπορίου των όπλων σε διεθνέ επίπεδο και εδώ θα αναφερθώ σε μερικά μόνο σημεία. Η και επιβάλλει σε όλα τα συμβαλόμενα μέρη να έχουν ένα σύστημα εθνικών ελέγχων με ένα κατάλογο που να μιλάει για τη μεταφορά όπλων. Εξαγωγές δηλαδή, εισαγωγές, transit, Οι χώρες επίσης πρέπει να κάνουν μια αξιολόγηση στις εξαγωγές όπλων τους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ένα σύστημα σαν και αυτό δηλαδή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1998 μέσω του κώδικα δεντολογίας που έχει. Το κείμενο προβλέπει ότι κάθε αξιολόγηση κινδύνου ε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο για την υγεία, και την παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς ε, δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να λαμβάνει υπόψη τρομοκρατικές πράξεις ή ε, το διεθνές ε, έγκλημα, μεταξύ άλλων. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται αφού ληφθούν υπόψη μέτρα άμβλυνσης των αρνητικών αυτών συνεπειών. Δεδομένης της συζήτησης που ακολούθησε, μπορούμε να πούμε ότι τελικά το εύρος εφαρμογής είναι αρκετά μεγάλο. Επιπλέον από ότι τα συμβατικά όπλα που περιλαμβάνονται στο Μητρό των ε, Ηνωμένων Εθνών υπάρχουν και τα ελαφρά όπλα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εδώ. Να υπογραμμίσουμε και τα πυρομαχικά και τα συστατικά όπλα που περιλαμβάνονται και αυτά. Παρ' όλα αυτά, το πεδίο εφαρμογή είναι ατελές γιατί δεν έχουμε ορισμό του όρου εξαγωγή. Οπότε φαίνεται ότι αποκλίνονται οι μεταφορές που μπορούν να είναι δώρα, εκχωρήσεις, μεταφορά τεχνολογίας, δάνεια κτλ. Οπότε Υπάρχει ακόμη και το θέμα συν, συμπερίληψης των ρομπότ ε, ή άλλων κατηγοριών όπλων που δεν περιλαμβάνονται. Επίσης, κάποιες διατάξεις ε, είναι σχετικά όριστες, κάτι που συμβάλλει στην ε, γενικότητα και την αφησιμία πολλών διατάξεων της συνθήκης. Για παράδειγμα, Έχουμε πολύ όριστες διατυπώσεις, όπου δει, όπου είναι δυνατό, όπου είναι κατάλληλο, ή οι χώρες ή ε, παροτρύνονται να. Αυτές οι αόριστες ε, διατυπώσεις ε, ανοίγουν το δρόμο για διαφορετική ερμηνεία και πρακτική, κάτι που αντιβαίνει στον οικουμενικό χαρακτήρα της συνθήκης. Επίσης, το κείμενο παρουσιάζει και κάποιες αδυναμίες. Θα αναφερθώ σε μία βασική που αφορά την έννοια του σημαντικού κινδύνου για την αξιολόγηση ε, τη δυνατότητα της δυνατότητας εξαγωγής. Φαίνεται ότι είναι υποκειμενικός αυτός ο χαρακτηρισμός. Ε, επίσης ε, γίνεται μια ιεράρχηση του κινδύνου από τον ίδιο τον εξαγωγέα. Και χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία και το Λίχτενστάιν ήδη έχουν εξαγγείλει κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνθήκης ότι θα ερμηνεύσουν τον κίνδυνο ως έκδηλο κίνδυνο, που είναι λιγότερο υποκειμενικός όρος από τον σημαντικό κίνδυνο που διακυβεύει άλλωστε τα κριτήρια αξιολόγησης ε, λόγω της υποκειμενικότητας. Το κείμενο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των μερών, αλλά τουλάχιστον βελτιώνει ε, τη γενικότερη ασφάλεια ενισχύοντας τον έλεγχο στη, στο Διεθνές Εμπόριο Όπλων. 115 χώρες ε, έχουν ήδη υπογράψει τη συνθήκη και 8 την έχουν κυρώσει. Οπότε απομένει το θέμα της εφαρμογής της συνθήκης αυτούσιας. Η οι χώρες μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε οι πρόοδες που έχει γίνει μέσω κάποιων διατάξεων να εφαρμοστούν αυστηρά και οι αδυναμίες του κειμένου να μην ε, αλλοιώσουν τη γενική εφαρμογή. Γι' αυτό και η διεθνή συνεργασία και συνδρομή θα είναι το καταλληλότερο μέσο για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική εφαρμογή. Βέβαια, μερικές χώρε δεν διαθέτουν εθνικό σύστημα ελέγχου. Άλλες χώρες έχουν μια ατελή νομοθεσία. Και εδώ περιλαμβάνω και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η κοινή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτεί από τα κράτη-μέλη να κάνουν κοινοποίηση των εισαγωγών τους. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ άλλες χώρες διαθέτουν παροχημένη νομοθεσία μερικές φορές που χρονολογείται από την ε, απεικιοκρατική εποχή. Θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Επίσης, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να τηρήσουν τη συνθήκη. Για πολλέ θα πρέπει να αλλάξει η εθνική νομοθεσία, να δημιουργηθούν αρμόδιες αρχές, να θεσπιστούν νέε διατάξει, να εκπονηθούν νέα έγγραφα, κάτι που προϋποθέτει ε, σημαντικούς ε, οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνδρομή. Βέβαια, τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν αρρωγή από τα κράτη-μέλη, από περιφερειακές οργανώσεις και από την κοινωνία των πολιτών. Ως περιφερειακή οργάνωση που διαθέτουμε συγκεκριμένες διατάξεις για το εμπόριο όπλων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ήδη να εντοπίσει κάποια στοιχεία της συνθήκης για τα οποία θα μπορούσε να παράσει συνδρομή και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη που το ζητούν. Επίσης, να θαρρύνει τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν στο ε, εθελοντικό ταμείο συνδρομής που προβλέπει η συνθήκη. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε, στο σημαντικό θέμα της ερμηνείας της συνθήκης. Γιατί υπάρχουν ανακρίβειες, ελλειπείς ορισμοί και αμφισημίες που δυστυχώς ε, αυξάνουν τον κίνδυνο διαφοροποιημένης ερμηνείας. Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας ε, υψηλός βαθμός κοινή ερμηνείας από τα κράτη-μέλη, ώστε να έχουμε αποτελεσματική, ολοκληρωμένη και συνεπή εφαρμογή των ε, διατάξεων της συνθήκης. Επίσης θα πρέπει να γίνει εσωτερισμός των πρακτικών γιατί εδώ και χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι η ερμηνεία των κριτηρίων δεν είναι πάντα εύκολη. Εντάξει, να έρθω στην ουσία. Θα πρέπει να ενισχυθούν τα κρατημέλη ώστε να υιοθετήσουμε μια κοινή ερμηνεία των διατάξεων της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να ενισχύσει την εφαρμογή και τη δέσμευση όλων των κρατών ε, μελών του ΟΗΕ με την ε, διοργάνωση σεμιναρίων και να προάγει όσο γίνεται την κοινή ερμηνεία των κριτηρίων της συνθήκης. Σας ευχαριστώ. Ωραία. Το κείμενο υπάρχει. Έδωσα το λόγο σε όσου το ζήτησαν οι ευρωβουλευτές τώρα. Ό,τι παρατηρήσεις έχουν να κάνουν είτε ακαδημαϊκού χαρακτήρα και διπλωματικού χαρακτήρα, όποιο έχει να κάνει άλλη παρατήρηση μπορεί να απευθυνθεί στους ευρωβουλευτές και οι τροπολογίες μέχρι 18 Δεκεμβρίου στι 5 το απόγευμα είναι η προθεσμία για την υποβολή τους. Για οτιδήποτε άλλο μπορείτε να τα συζητήσετε εκτός, αλλά εδώ ό,τι υπόθηκε υπόθηκε. Και για τις δύο και για τα δύο σημεία, και για την γνωμοδότηση του κύριου Λίσεκ και για το δικό μου σχέδιο ψηφίσματος ισχύ προθεσμία που σας έδωσα πριν για την υποβολή τροπολογιών. Θέλουμε το Φεβρουάριο να περάσει στην Ολομέλεια ε, το θέμα αυτό με συζήτηση ε, στην Ολομέλεια και νομίζουμε ότι και είπα το εκπρόσωπος θα είναι παρούσα τότε. Αυτά για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ και έληξε η συνεδρίασή μας.